Σε μερικά λεπτά θα ξαναρχίσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ όμως εντωμεταξύ τους συναδέλφους είτε να αποχωρήσουν γρήγορα και ήσυχα είτε να ξανακαθίσουν στις θέσεις τους. Μερικά δευτερόλεπτα διακοπή.